Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να σας καλησπερίσω και σαν ε, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με, την, ε, με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής θα ήθελα να καλωσορίσω όλους σας σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της ΔΚΑΜ και της ΔΙΛΑΤ να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του στον συμπρόεδρο της συνάντησης, τον κύριο Χουαρέβη, πρόεδρο της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και τον αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κεντρική Αμερική, κύριο Γκαμπριέλ Μάτο. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους επισκέπτες μας, τον κύριο Μαρτινέθ, Υπουργό Εξωτερικών του Ελ Σαλβαδόρ, τον κύριο Ασμπούν, Γραμματέα για την Διακυβέρνηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ, τον κύριο Μοράλες, αναπληρωτή γραμματέα για τη διακυβέρνηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας του Ελσαλβαδόρ, τον κύριο Τσάβες Μένα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια του Πολίτη, τον κύριο Κατεϊάνος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια του Πολίτη επίσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω και όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών και ιδίως τον κύριο Εσκαλάντε Ασμπούν, επιτετραμένο της Πρεσβείας του Ελσαλβαδόρ. Να καλωσορίσω επίσης και όλους τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντελαρίτσια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και να σας πληροφορήσω για πολλοστή φορά βεβαίως ότι η διερμηνία παρέχεται στις, ε, στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα γαλλικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ελληνικά και στα ιταλικά. Και επίση να σα ενημερώσω στο σημείο αυτό ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Το σχέδιο της ημερήσια διάταξη, κύριοι συνάδελφοι, το έχετε, σας έχει διανυμηθεί στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά, γερμανικά και ελληνικά και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, η ημερήσια διάταξη θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί. Πριν δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο αυτή τη συνάντηση, τον κύριο Χαρέβη, επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια εξ ονόματο τη αντιπροσωπεία τη ΔΕΚΑΜ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον, στο, Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κύριο Μαρτινέ για να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλεια του Ελ Σαλβαδόρ. Η αντιπροσωπεία μα, όπω ξέρετε, έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία και προσοχή στο πρόβλημα τη ασφάλεια των πολιτών στην Κεντρική Αμερική ένα θέμα προτεραιότητας της χώρας του λεγόμενου Βορείου Τριγώνου, που είναι μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτηνιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και η κοινή γνώμη στην περιοχή πιστεύουν ότι η εκτεταμένη εγκληματικότητα, τα υψηλά ποσοτά της θανατηφόρας βίας και η συνολική υποβάθμιση της ασφάλειας του πολίτη είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της Κεντρικής Αμερικής για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών. Στις 30 Ιουλίου του 2014, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε μια στρατηγική για την ασφάλεια των πολιτών στην Κεντρική Αμερική και στην Καραϊβική, την οποία ακολούθησε ένα σχέδιο δράσης το 2015. Οι κατευθύνσεις που προτάθηκαν των δράσεων αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, η οικοδόμηση μιας κοινωνικής πολιτικής ατζέντας για την ασφάλεια των πολιτών, η ενίσχυση της ικανότητας των κυβερνήσεων να παρέχουν ποιοτικέ δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η, η αντιπροσωπεία μας συζήτησε την ασφάλεια των πολιτών σε διάφορες περιπτώσεις στι συναντήσει μας και φυσικά κατά τι επισκέψει μας σε χώρε Κεντρική Αμερικής και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να ακούσουμε από πρώτο χέρι σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στο Ελ Σαλβαδόρ αλλά και το βαθμό στήριξη που παρέχεται στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν σταματήσω εδώ, θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ότι η αντιπροσωπεία μας σχεδιάζει να επισκεφθεί τη χώρα σας τον επόμενο χρόνο και ελπίζω και ότι θα έχουμε την ευκαιρία τότε να δώσουμε συνέχεια στη σημερινή συνάντηση και να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τα όσα θα συζητήσουμε σήμερα και αφορούν στην, ε, ε, στην βελτίωση της ασφάλειας της χώρας σας. Ε, με αυτή την ευκαιρία λοιπόν σας δίνω και το λόγο να ξεκινήσει η κουβέντα μας. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Bien, muchísimas gracias. Eh, muy... Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς τους ε, ευρωβουλευτές ε, και κυρίως τους πρόεδρους των επιτροπών και όλους ιδιαιτέρως ε, στην Επιτροπή για την Κεντρική Αμερική. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας αφιερώνετε αυτό το χρόνο, το χρόνο σας για να σας παρουσιάσουμε τη στρατηγική ασφάλεια στο Ελσαλβαντόρ που ευτυχώς ήδη έχει αποφέρει σημαντικούς καρπούς, ήδη έχει παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα, ώστε να αλλάξει επιτέλους αυτή η ιδέα που υπερίσχε μέχρι τώρα, ότι το, το Ελσαλβαδόρ και οι χώρες ε, του Βορείου Τριγώνου είναι πολύ επικίνδυνες. Και αν ε, διαβάσετε πρόσφατες ειδήσει από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, και όπως θα διαπιστώσετε και από την παρουσίασή μας, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 65% τις ανθρωποκτονίες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο φέτος, σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016. Και μάλιστα αυτή η τάση έχει αρχίσει και ατρεώνεται πια από πέρσι τον Απρίλιο με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης Σίγουρο Ελσαλβαδόρ Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σφαιρικό σχέδιο που περιλαμβάνει και συνιστώσει πρόληψη, συνιστώσει φυσικά δίωξη ε, των ε, αξιόπινων πράξεων, αλλά και συνιστός ε, προστασίας, αποκατάστασης, επανένταξης, συνδρομή και προστασίας των θυμάτων και θεσμικής ενδυνάμωσης των διαφόρων τομέων του σχεδίου αυτού για το σίγουρο, το πιο το ασφαλέστερο Ελσαλβαδόρ. Η εμπειρία αυτή ε, απορρέει από μια συμμετοχική διαδικασία. Γι' αυτό έχουμε εδώ και τον πρώην σύμβουλο Τσάβελς ε, από την ε, σύνυπαρξη του πολίτη και τον επιχειρηματία Ραφαέλ Καστεγιάνος που μαζί με εκπροσώπους των πανεπιστημίων, των πολιτικών κομμάτων, του επιχειρηματικού κλάδου, της κοινωνίας των πολιτών έλαβαν μέρος στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Και επίσης ε, συμμετείχαν σε αυτό και εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας. Ε, είχαμε χθε και την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το Συμβούλιο. Έχουμε τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης λαμβάνει μέρος στην σε αυτή και τον πρέσβη του Ελσαλβαδόρ και συμμετείχε και στο Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι από οργανώσεις Αμερικανικών κρατών και είχαμε και στο Συμβούλιο και άλλους εκπροσώπους χωρών που έχουν διαπιστευμένους πρέσβεις στο Ελσαρβαδόρ. Θέλουμε λοιπόν να μοιραστούμε μαζί σε αυτή την εμπειρία που εστιάζεται φυσικά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι και ο ακρογωνιαίος λήθος της δημοκρατικής κοινο... κοινωνίας που δημιουργήθηκε μετά τη σύναψη των Ελληνευτικών συμφωνιών στο Ελσαλβαδόρ. Και είναι σημαντικό να βρεθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ της εκτέλεσης ενός αποτελεσματικού σχεδίου που μας επιτρέπει σημαντική θεματική μείωση του επίπεδου των ανθρωποκτονιών και ταυτόχρονα να συνδυάζουμε αυτή την προστασία με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι η σημαντική δέσμευση της ε, σημερινή κυβέρνηση που απορρέει και από τις ε, ειρηνευτικέ συμφωνίε που έχουμε συνάψει. Αυτά. Ο κύριος Άτο Ασμπούν, που είναι γραμματέας ε, περί διακυβέρνησης θα κάνει την παρουσίαση με το PowerPoint. Και επίσης θα ήθελα να δώσουμε το λόγο και σε μέλη του Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου, για κάποια σύντομα σχόλια. Και μετά θα περάσουμε στο πιο σημαντικό σημείο που είναι οι δικές σας απορίες, ανησυχίες, προτάσεις, σχόλια, γιατί φαντάζομαι ότι θα δημιουργηθούν κάποιες ανησυχίες για επιπλέον θέματα του Εθνικού Συμβουλίου. Αλλά ήθελα σήμερα να επικεντρωθούμε κυρίως στα ζητήματα που άπτονται αυτού του Συμβουλίου. Αυτά θερμά ευχαριστώ και χωρίς ε, άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον γραμματέα περί διακυβέρνησης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> αγαπητέ Πρωθυπουργέ Μαρτίνες. <clears throat> Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους παρόντες, τους ευρωβουλευτές, Υπουργέ Εξωτερικών, συγγνώμη, και να τους ε, θα ήθελα να χαιρετήσω και τον εξοχότατο πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, τον κ. Σεγούρα, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ χωρίς την βοήθειά του και όπως είπε και ο υπουργό Εξωτερικών μας, η παρουσία του στην χώρα μας είναι, όπως είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της εκπροσώψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Θα περάσω τώρα λοιπόν στο, στην ε, παρουσίαση των ε, εκπροσώπων μας από το Συμβούλιο Διακυβέρνηση, ο κ. Κασταγιάν και ο κ. Μένα. Το Συμβούλιο Ασφάλειας, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Πολιτών στο Σαλβαδόρ, στον Σαλβαδόρ, είναι μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, είναι ένας φορέας συνεννόησης, επίτευξης συμφωνίας, για ένα θέμα το οποίο είναι κεφαλαίο για τους πολίτες και είναι το θέμα της ανασφάλειας των πολιτών. Δεν είναι μόνο το θέμα της εγκληματικότητας. Είναι το πρόβλημα της ανασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες εάν το δούμε σε συνολικό τρόπο. Δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο προέρχεται από πολλές αιτίες, από πολλά φαινόμενα. Γι' αυτό εμείς έχουμε εκπονήσει μια συμπεφωνημένη και συντονισμένη πρόταση για αυτό το σχέδιο ασφάλειας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί τομείς τη ε, κοινωνία μας οι οποίοι ενεπλάξαν στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου που είναι ένα συνενετικό σχέδιο. Υπήρξαν διάφορα στρώματα, διάφοροι φορεί της κοινωνίας μας που θέλησαν να δημιουργήσουν μια κρατική πολιτική για τα θέματα ασφάλεια στο Ελσαλβαδόρ, ώστε να μπορέσει ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση στη χώρα μας, να συνεχίσει η υλοποίηση αυτού του σχεδίου γιατί ξέρουμε ότι έχει εμπλέξει όλους αυτούς τους τομείς οι οποίοι συμμετέσχουν στην ε, εκπόνηση και επεξεργασία αυτού του σχεδίου. Πρόκειται λοιπόν για φορείς οι οποίοι συμμετέχουν <clears throat> στον κρατικό μηχανισμό. Είναι σημαντική η παρουσία των τοπικών αρχών αυτοδίκησης και φυσικά δεν χρειάζεται εδώ να πω περισσότερα για να τονίσω πόσο σημαντική είναι η παρουσία των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινοτήτων. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Επίσης υπάρχουν εκπρόσωποι των εκκλησιών, της Καθολικής Εκκλησίας και των ιστορικών δογμάτων στο Ελσαλβαδόρ και αυτοί είναι παρόντες στον με τους φορείς τους και εργάζονται άμεσα στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, τα μέσα ενημέρωσης, οι οργανώσεις των εργοδοτών, τα πολιτικά κόμματα, άτομα τα οποία έχουν ειδικέ ε, ικανότητες και προσόντα για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ε, ασφάλειας των πολιτών. Έχουν τη δυνατότητα ως εμπειρογνώμονες λοιπόν να συνεισφέρουν προτάσεις για το θέμα αυτό <clears throat> και όπως έλεγε και ο υπουργό μας υπάρχουν και εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας. Σας <clears throat> τόνισα προηγουμένως ότι μία από τις σημαντικές μας επιτεύξεις είναι ότι πρόκειται για μια πολιτική της κυβέρνησης αλλά που βασίζεται στην συνένεση. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εγώ πρέπει να αποδεχτώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία συμμετείχα εγώ είχαν με κάνει το λάθος να ζητήσουμε από τους ε, φορείς της κοινωνίας να συμμετάσχουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου. Αλλά μας είπαν γιατί να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια συζήτηση αν μετά δεν θα εμπλακούμε στην εκπόνηση του συνολικού σχεδίου και θα διαβουλευτούμε απλώς. Οπότε οδηγηθήκαμε στο να έχουμε μια κοινή εκπόνηση του σχεδίου αυτού, να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες από κοινού και με πόρους που προέρχονται από ίδιους πόρους. Υπάρχει φυσικά μια συνεισφορά από την κυβέρνηση για την ε, υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ένα άλλο σημείο στο οποίο είχαμε σημαντικές ε, <clears throat> πρόοδους ήταν ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όπως είπε ο Υπουργός εξωτερικός μας αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον μόνιμο και αυστηρό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μην επιτρέψουμε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ειρήνευσης, που ήταν η δημιουργία της Εθνικής Αστυνομίας και επίσης και άλλες πτυχές της ε, συμφωνίας αυτής που έχουν να κάνουν με την πάταξη της εγκληματικότητας. Μπορώ να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που είναι επικεφαλής αυτού ο, ο κύριος Μαρτίνες για να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος και να εξασφαλιστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω αυτού του αστυνομικού φορέα. <clears throat> Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει συνέχεια να αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας ένα αένα, ένα διαρκή αγώνα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων του πληθυσμού μας. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για την κοινή δράση μεταξύ της ε, αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις δρούν με τον έλεγχο και υπό την ηγεσία της Εθνικής Αστυνομικής Αρχής και πάντα στον, στο πλαίσιο του σεβασμού των κανονισμών που προκύπτουν από το σχέδιο για το ασφαλές Σαλβαδόρο. Όπως έλεγα επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να σας αναφέρω είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό σημείο της ε, εφαρμογής του σχεδίου το Ασφαλές Σαλβαδόρ και επίσης σας τονίζω ότι εργαζόμαστε με δικούς μας πόρους για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Κάτι ακόμα το οποίο δεν αναφέρεται στην ε, παρουσίασή μου, αλλά είναι σημαντικό, είναι ο τρόπος με τον οποίο συναρθρώνονται οι διάφορες εθνικές αρχές, δηλαδή η εισαγγελική αρχή, το ανώτατο δικαστήριο και άλλες εθνικές αρχές οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Έχει πέντε βασικούς άξονες στο πρόγραμμα ε, ασφαλές Σαλβαδόρ με 133 επιμέρους δράσεις και προβλέπεται σε πέντε χρόνια να αφιερωθούν σε αυτό 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Κύριος άξονας είναι η πρόληψη της βίας. Εδώ για τα πέντε χρόνια θα δοθούν 1,55 δισεκατομμύρια. Και κυρίως εδώ μας ενδιαφέρει <clears throat> η δημιουργία απασχόλησης για τους νέους. 33% από αυτές τις θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να αφορούν γυναίκες. Επομένως, η πρόληψη της βίας είναι ο βασικός άξονας του προγραμματός μας, του σχεδίου <clears throat> το Ασφαλές Ελσαλβαδόν. γιατί προσπαθούμε να εξαλείψουμε μία από τις κύριες αιτίες εγκληματικότητας που είναι η ανεργία. Οι γνώστες του σχεδίου γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό σε χώρες όπως το Ελσαλβαδό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση. Δεύτερη πτυχή είναι η ανεργια οι γνωστες του σχεδιου γνωριζουν πολυ καλα οτι αυτο σε χωρες οπως το ελσαρβαδο ειναι μια παρα πολυ σημαντικη προκληση δευτερη πτυχη ειναι η διωξη και η πάταξη του εγκλήματος με 155 εκατομμύρια προϋπολογισμό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Επομένως εδώ πρόκειται για ενέργειες που γνωρίζουν όλοι ως καταστολή της εγκληματικότητας και έλεγχος των ποινικών διαδικασιών. Τρίτο στοιχείο είναι η αποκατάσταση και επανενσωμάτωση με 180 εκατομμύρια. Τέταρτον είναι η προστασία και η μέρημνα για τα θύματα της εγκληματικότητας με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων και επίσης έχουμε την θεσμική ενίσχυση με χρηματοδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ δολαρίων. Η τρίτη πτυχή που περιλαμβάνεται στο σχέδιο το ασφαλές El Salvador είναι μια στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Εμείς εστιάζουμε τις ε, διοκτικές δυνάμεις και τους πόρους στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει το κυριότερο, τα κυριότερα προβλήματα εγκληματικότητος. Και φυσικά αυτά τα σημεία εγκληματικότητος διασταυρώνονται με τον χάρτη της ένδυας. Έχουμε 261 δήμους, 50 δήμοι είναι αυτοί όπου συγκεντρώνεται σχεδόν πλήρως το πρόβλημα της ε, βίας και της εγκληματικότητας. Και βλέπετε εδώ ότι πράγματι αντιστοιχούν όλα αυτά τα περιστατικά εγκληματικότητας με τις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη ένδια. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε καταρχήν με το να εστιάσουμε την προσοχή μας σε δέκα δήμους όπου είναι πιο έντονο το πρόβλημα θα προχωρήσουμε στους 27 ε, και μετά θα φτάσουμε στους 50 δήμους ώστε έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Όπως είπε ο κύριος Μαρτίνε, μία από τις επιτυχίες που έχουμε καταγάγει βάσει των ενδεικτών μας είναι ότι έχει μειωθεί σημαντικά η εγκληματικότητα. Στην πράξη είναι 62% η μείωση των ανθρωποκτονιών στη χώρα μας βάσει των στοιχείων που έχουμε συλλέξει. γιατί στο Ελσαλβαδόρ αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται θετικά. Έχουμε λοιπόν και ένα σημαντικό ενδείκτη ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση στη μείωση του αριθμού των ε, ανθρωποκτονιών. Είναι μη αντιστρεπτή αυτή η μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών. Έχουμε μπει λοιπόν σε αυτό το δρόμο εδώ και πολύ καιρό για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ε, ανθρωποκτονίες και με τους ε, δείκτες μας μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η τάση η οποία διαγράφεται δεν είναι συγκυριακή αλλά είναι πραγματική, είναι μόνιμη. Γι' αυτό είναι σημαντική η επένδυση η οποία έχει γίνει στους Δήμους, που είναι η δήμη όπου επικεντρώνεται περισσότερο <clears throat> η, η βία και οι ανθρωποκτονίες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς <clears throat> δράσεις, οι οποίες όμως θα ξεκινούν από την τοπική κοινότητα. Δεν θα είναι οι αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες θα ε, παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά οι τοπικές κοινότητες. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και για την παροχή των ε, πόρων που δόθηκαν για τις επενδύσεις αυτές σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα της ε, πρόληψης. Ένα άλλο σημείο που θέλω να θίξω είναι η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου. Υπάρχει ένας ειδικό φόρος για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ο φόρος εισοδήματος για τους ε, αυτός με υψηλό εισόδημα που αποδίδει περίπου 110 εκατομμύρια ε, δολάρια το 2017 και περίπου 500 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. 5% φόρος επί των περιουσιών που δημιουργούν εισόδημα πάνω από 500.000 ετησίως και επίσης ε, φόρος στις τηλεπικοινωνίες. Δεύτερη πτυχή της χρηματοδότησης είναι η διεθνή συνεργασία και ο δανεισμός, περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 25 έχουν ήδη εγκριθεί. Τρίτο στοιχείο είναι ο εθνικός προϋπολογισμός και οι δημοτικοί προϋπολογισμοί, περίπου 500 εκατομμύρια σε 5 χρόνια <clears throat> και επίσης συμμετοχή τοπικών και διεθνών ιδρυμάτων, περίπου 100 εκατομμύρια στα επόμενα 5 χρόνια. Αυτές λοιπόν είναι οι χρηματοδοτικές πτυχές για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου. Έχουμε και μία σειρά από συμπληρωματικά σχέδια και προσπάθειες <clears throat> για να δημιουργήσουμε ένα πιο έφορο κλίμα για την ε, μείωση της εγκληματικότητας είναι κυρίως ενέργειες εκπαιδευτικού χαρακτήρα και κοινωνικού χαρακτήρα. Το ποινικό σύστημα στο Ελσαλβαδόρ είχε καταρρεύσει το παρελθόν. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε προγράμματα τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι γίνεται πραγματική αποκατάσταση και επανενσωμάτωση των ατόμων που έχουν περάσει στην εγκληματικότητα. Και υπάρχει επίσης και πρόγραμμα για την μέρημνα και την προστασία των θυμάτων της ε, βίας. Έχουμε με τα τοπικά συστήματα λοιπόν αυξήσει την προστασία σε αυτά τα άτομα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό πρόγραμμα είναι η παροχή θέσεων απασχόλησης και η δημιουργία απασχολησιμότητας για τους νέους. Έχουμε ήδη χίλιους νέους οι οποίοι είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε την επανενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα Εργαζόμαστε λοιπόν για να ξαναφέρουμε αυτά τα παιδιά, <clears throat> τους νέους και τις νέες που έχουν εξέλθει από το σχολικό σύστημα, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στο σύστημα αυτό. Και τέλος φυσικά έχουμε και ενέργειες στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπου έχουν ε, επωφεληθεί περίπου 250.000 νέοι από όλα αυτά. Και βλέπετε εδώ πέρα στο γράφημα, δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που σας είπα, γιατί τα ανέφερα προηγουμένως. Βλέπετε αυτό το γράφημα το οποίο παρουσιάζει την ε, τάση στις ε, ανθρωποκτονίες, τον αριθμό των ανθρωποκτονιών για κάθε 100.000 πολίτες από το 1980 ως το 2016. Ο δόκτωρ Τσάβεσμενα Μένα μας έχει δώσει αυτό το γράφημα και βλέπετε πως έχει μειωθεί ο αριθμός αυτών των ανθρωποκτηνωνιών και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια ουσιαστική μείωση. Έχουμε μια σταθερή λοιπόν μείωση. Και εδώ βλέπετε λοιπόν και από το γράφημα το επόμενο γράφημα πως η συγκέντρωση των πόρων, δηλαδή η δημιουργία προτεραιοτήτων στις πιο επικίνδυνες περιοχές όπως προβλέπει το σχέδιο επέτρεψε να υπάρξει μια σταθερή μείωση των ανθρωποκτονιών στους 10 δήμους όπου δώσαμε πρώτη προτεραιότητα. Είχαμε λοιπόν 430 λιγότερες ανθρωποκτονίες το 2016 σε σχέση με το 2015 με επομένω μείωση 25%. Και φυσικά υπάρχουν και δήμοι όπου ε, στο παρελθόν δεν υπήρχαν καθόλου ανθρωποκτονίες, όπου υπήρξε μια αναζωοπήρωσή τους. Όλα αυτά εγγράφονται λοιπόν στο γενικό σχέδιο για τον αγώνα κατά της ανασφάλειας. Έχουμε και άλλα δύο σχέδια για, το... για την εκπαίδευση στο Σαλβαδό για να υπάρξει αλ... αλφαβητισμός σε όλους και εκπαίδευση και υπάρχει και το Συμβούλιο Αηφορίας το οποίο επίσης λειτουργεί επί τη βάση μιας συμφωνίας σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού περιβαλλοντικου ιστού. Προσπαθούμε λοιπόν με όλους αυτούς τους τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι η συμφωνία ε, και η συνένεση στο Σαλβαδόρ θα παραμείνει μια πολιτική που θα είναι η πολιτική του κράτους μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έχει ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τώρα για την σύναψη μιας δεύτερης γενιάς συμφωνιών, ε, δεύτερης γενιάς μετά από την πρώτη συμφωνία που υπεγράφει το 1992 στο τέλος του ε, εμφυλίου πολέμου που έλαβε χώρα στη χώρα μας κυρίως τη δεκαετία του 1980, θεωρούμε ότι μετά από αυτή την πρώτη γενιά συμφωνιών μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, χρειαζόμαστε τώρα να περάσουμε σε μια δεύτερη φάση. Και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα από τα βασικά προβλήματα της χώρας μας, το θέμα της άκρας ένδυας και υπάρχει η επεξεργασία του σχεδίου αυτού με την παρουσία και του Υπουργείου Εξωτερικών και με την παρουσία διαφόρων φορέων της κοινωνίας μας για να εξασφαλίσουμε τη σύναψη μιας δεύτερης συμφωνίας η οποία θα είναι απαράγραπτη για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και που θα πρέπει να αποτελέσει την κρατική πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν προκύπτουν από την συμφωνία αυτή για το ασφαλές Ελσαλβαδόρ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, θα ήθελε θα ήθελαν οι, κυρία, η κύριοι Καστεγιάνος και Τσάβες Μένα να συμπληρώσουν την παρουσίαση για το σχέδιο ασφαλείας για το Ελσαλβαντόρ. Αλλά παρακαλώ εν συντομία για να έχουμε κάποιο χρόνο για τη συζήτηση να μας εκφράσετε και τις απορίες και τις ε, παρατηρήσεις σας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή, τους Ευρωβουλευτές, τον συνάδελφο και πρέσβη Χαούμε Σεγούρα για τη δεράστια προσπάθεια που έχει κατεβάλει. Μας έχετε βοηθήσει τα μάλα και με κονδύλια που πραγματικά έχουν πιάσει τόπο. Σας διαβεβαιώ ότι τα χρήματά σας ε, έχουν πιάσει τόπο. Εγώ ανήκω στην αντιπροσωπεία, επιχειρηματίας, αλλά και δημοσιογράφος ταυτόχρονα, ε, γιατί γράφω σε περιοδικά. Ε, φυσικά είμαι σε διαφορετική ιδεολογική παράταξη από την κυβέρνηση και έτσι αυτό είναι έμπρακτη απόδειξη ότι ο τρόπος που δουλεύουμε δεν ε, ε, τυφλώνεται από ιδεολογίες, αλλά βασικό μας μέλημα είναι το συμφέρον της χώρας. Συμμετέχω λοιπόν στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας μετά από πρόταση του παιδικού μου φίλου, του Άτο Ασμπούν, και μάλιστα από την αρχή τη ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου, με αρκετέ αμφιβολίε, γιατί μια κυβέρνηση τη αριστερά που οι φίλοι μου έλεγαν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ε, μου, με προειδοποίησαν οι φίλοι μου ότι θα σε χρησιμοποιήσει η αριστερή κυβέρνηση. Είπα όμως καλύτερα να με χρησιμοποιήσει και καλύτερα να κάνω λάθος δίνοντας μάχη παρά να αρκούμε να ασκώ επικρίσεις ε, ε, από την ασφάλεια του καναπέ μου ή σε δεξιώσεις πίνοντας ένα ποτήρι κρασί. Γι' αυτό ήθελα εμπράκτως να συμμετέχω στην παρουσίαση και στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Και μάλιστα έχω και ένα σημαντικό ε, σχέδιο 300 ε, εκταρίων για τη δημιουργία ενός ε, γηπέδου γκολφ. Έχουμε και πολλούς αποσχολούμενους 200 με 300 στο σχέδιο αυτό. Και μάλιστα, την... μάλιστα γύρω από το σχέδιο αυτό, το, γήπεδο γκολφ που έχουμε κάνει, υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλοί βάλτοι και και ένας ε, νεαρός, 23χρονος, 24χρονος, ένας πολύ ε, νέος, ε, με δύο παιδιά, η γυναίκα του επίση εργαζόμενη, κλασική φτωχή οικογένεια που πηγαίνει στις 8 το βράδυ ε, να συναντήσει τη γυναίκα του στη, που βγαίνει από το λεωφορείο και μάλιστα έχει συμμορίες, έχουμε πολλές συμμορίες γύρω από εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνη η περιοχή γύρω από το γήπεδο και πρόσφατα είχαμε και μια ανθρωποκτονία και αυτό θέλουμε να σταματήσουν, να σταματήσουν αυτές οι, οι ανθρωποκτονίες αυτές τις επικίνδυνες περιοχές. Και μάλιστα πολλοί ε, κάτοικοι του Σαλβαδόρ, νέοι, θέλουν να αποδημήσουν γιατί δεν βλέπουν ελπίδα στη χώρα τους. Θέλουμε λοιπόν αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και αυτή η κατάσταση οφείλεται πρώτον λόγω της βίας, αλλά και δεύτερον επειδή ως κοινωνία δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετές θέσεις απασχόλησης για να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτούς τους νέους. Κάθε χρόνο έχουμε 50.000 νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας αλλά δεν βρίσκουν, είναι μάλλον να έχουν, θα μπορούσαν να ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν έχουν θέσεις για να απασχοληθούν. Και μάλιστα ε, τρία εκατομμύρια συμπολίτε μας ε, μένουν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε μεγάλο απόδημο ε, τμήμα του πληθυσμού μας. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και εγώ δεν είμαι από το κατεστημένο, έρχομαι απ' έξω, παρόλο που έχουμε γίνει φίλοι μεταξύ μας και σας διαβεβαιώ ότι αυτό το σχέδιο λειτουργεί και είμαι ζωντανό παράδειγμα και τη απόδειξη της αποτελεσματικότητας αυτού του σχεδίου. Και το αν κάποιος θέλει να συμμετέχει ε, στα τεκτενόμενα θα πρέπει να λαμβάνει μέρος στο διάλογο, στις συζητήσεις και μπορεί να μην ήταν εύκολο όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι με το ρεαλισμό τα καταφέραμε. Και θα ήθελα να καταθέσω και εγώ τη μαρτυρία μου ότι τα πράγματα έχουν μπει στο αυλάκι και αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία θα δημιουργήσουμε ένα πολύ θετικό προηγούμενο για όλο τον κόσμο και θα γίνουμε στο Ελ Σαλβαδόρ υπόδειγμα προς για την παγκόσμια κοινότητα. Βέβαια, είχαμε τον πρώτο χρόνο πολλά θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει εξίσου καλά αποτελέσματα να έχουμε και για την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω να εκφράσω μάλλον την ευχαρίστησή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο. Όπως θα θυμάστε, το Σαλβαδόρ ε, πέρασε έναν εμφύλιο πόλεμο που δίρκησε πολλά χρόνια στη δεκαετία του 1980. Και βεβαίως τότε επικράτησε βία. Σε αυτή τη μεταπολεμική περίοδο, από το 1990 25 χρόνια δηλαδή μεταπολεμική περίοδο, τα πρώτα χρόνια χαρακτηρίστηκαν ε, από αύξηση της βίας. και αυξήθηκε μέχρι και 170% ε, τα πρώτα 10-12 χρόνια. Στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή μείωση και μετά πάλι αυξήθηκε ακόμα 30%. Όλα αυτά μέσα σε ένα πλέγμα πολιτικών που βασικά είχαν προσανατολισμό την καταστολή του εγκλήματος Και με βάση τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας, ε, στην, οποία, στην, στην εκπόνηση της οποίας συμμετείχα και εγώ, από το 2010 και στη συνέχεια υπήρξε μια τάση μείωσης ε, των ανθρωποκτονιών ε, ανά 100.000 κατοίκους και κυρίως με την εφαρμογή και την εκτέλεση του σχεδίου για το ασφαλέ Σαλβαδόρ που εξηγήσαν ε, οι δύο κύριοι μιλητέ και η τάση είναι πολύ σαφής. Και όπως είπε ο Υπουργό Ιστορικών Μαρτίνεθ, από πέρυσι μέχρι φέτο στην ίδια ημερομηνία ε, καταφέραμε μείωση 65%. Και αυτό ε, οφείλεται στο ότι είναι ένα καθολικό, ένα σφαιρικό σχέδιο, ένα πλάνο ε, μέσα στο πλαίσιο του οποίου η έμφαση δίνεται στην πολιτική πρόληψης. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό Ε, όταν στηριχθεί περισσότερο η πολιτική πρόληψη, αυτό ακριβώς οδηγεί στην μείωση μάλλον στην διατήρηση αυτή της τάσης και στην μείωση της βίας στο Ελσαλβαδόρ. Και έπειτα θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει διάρκεια, χρονική διάρκεια. Η συμφωνία η ειρήνευσης ε, που γράφηκε στο τέλος του εμφυλίου πολέμου στην ουσία έδωσε την εξουσία στην ε, δεξιά στο Ελσαλβαδόρο που ακολούθησε πολιτικές ανάπτυξης αλλά ανάπτυξης με ε, μονόπλευρης οδηγώντας έναν κύκλο όχι ενάρετο ε, έτσι τελείωσε κάπως όμως υπό το πολιτικό χάσμα, ενώ το κοινωνικό χάσμα ξεκολουθεί να υπάρχει το πρέπει να προσπαθήσουμε προχωρώντας να καλύπτουμε ε, το κενό αυτό και να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε τις τα δευτικά αίτια της βίας στο Ελ Ήθελα και αυτό, αυτή την άποψη να την τονίσω και επίσης ε, να υπογραμμίσω ότι ως μέλος αυτής της, αυτού του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μπόρεσα να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στον σχηματισμό αυτής της ε, κρατικής πολιτικής που ήταν αποτέλεσμα μιας συνένεσης, συνένεσης άνευ προηγουμένου στο Ελσαλβαδόρ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψατε μου να απευθυνθώ στους προσκεκλημένους και σε όλους τους ε, συναδέλφους. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών του Ελσαλβαδόρου και όλη σας την ομάδα που είστε σήμερα εδώ παρόντες σε αυτή την μεικτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας για την Κεντρική Αμερική της οποίας προεδρεύει η φίλη μου Σοφία και της Αντιπροσωπείας Ερολάτ. Θα δώσω αμέσω τώρα το λόγο στους διάφορους ε, βουλευτές που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, σχόλια σε σχέση με αυτή τη σημαντική παρουσίαση. Θα ήθελα μάλιστα να σας πω αρχικά ότι εμείς βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Κεντρικής Αμερικής με πολύ μεγάλη στοργία, αγαπητέ Υπουργέ, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθούν προβλήματα τόσο μαζικής βίας που υπάρχουν σε ορισμένε από τι χώρε σα. Εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειές σας. Πολλέ φορές βλέπουμε χώρες όπως η δική σα, χωρίς να καταλαβαίνουμε καλά πόσο τεράστιο είναι το σύνολο των παραγόντων που οδηγούν σε αυτή τη τόσο γενικευμένη βία. Όταν για παράδειγμα κανείς ε, θυμηθεί όπως έλεγε και ο σύμβουλος εδώ ότι ο, ο πόλεμος δημιουργεί μια κουλτούρα βίας και η ζωή έχει μικρότερη αξία. Στις ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν δεν μπορούμε εύκολα να, να εκτιμήσουμε, να νιώσουμε πώς αυτές οι χώρες που υποφέρουν ε, επίσης και από φρικτή φτώχεια, πολλοί νέοι χωρίς κανέναν ορίζοντα, πολλές ε, απελάσεις από τη ΣΥΠΑ, ε, οργανωμένες ε, εγκληματικέ ομάδες που στην ουσία λειτουργούν ως παράλληλο κράτος, ε, μπορεί ναρκωτικών, τεράστια προβλήματα που δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το κρίνει ως αδυναμία ενός κράτους ή της δημοκρατίας στις χώρες αυτές. Είναι η συνέπεια μιας πραγματικά πολύ περίπλοκης πραγματικοτητα που απαιτεί τη στενή μα συνεργασία. Και γι' αυτό και πραγματικά η Ευρώπη έχει τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας, αναπτυξιακό πρόγραμμα και βοηθά όλες αυτές τις χώρες ε, στο πλαίσιο των συμφωνιών μας με την Κεντρική Αμερική αλλά και με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε. Θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι και ακόμη περισσότερο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές από την άποψη την γεωπολιτική για την ε, Λατινική Αμερική. Θέλουμε να είμαστε φίλοι της Λατινικής Αμερικής. Θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι της Λατινικής Λατινικής Αμερικής. Ε, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά κοινά ε, σημεία και μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί, αγαπητέ Υπουργέ. Και αυτό είναι το πνεύμα που μας συγκεντρώνει εδώ σήμερα και το πνεύμα που σίγουρα θα επικρατήσει στη διάρκεια των παρεμβάσεων των ε, συναδέλφων. Και άρα μετά την έγκριση και τη σοφία θα δώσουμε το λόγο στους και στις βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε ήδη έναν κατάλογο. Ωραία. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Λουίς Δεγκράντες έχει ζητήσει τον λόγο που είναι και πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την κυρία του ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Ε, αγαπητοί ε, προσκαλεσμένοι, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών του Ελσαλβαδόρ και απευθύνομαι και στους συνοδεύοντες τον κύριο Υπουργό και τον ε, επιχειρηματία που καταδεικνύει την ε, ευρεία συνένεση που ισχύει στο Ελσαλβαδόρ αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική υποχρέωση από όλους μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και να βρούμε μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Εγώ είχα την ευκαιρία στο παρελθόν να είμαι στη χώρα σας όταν ακόμα σοβούσε ο εμφύλος πόλεμος. Ήταν ο Ναπολεόν Ντουάρντε, ο οποίος είχε τότε την εξουσία, φίλος μου. Ήταν ο Φελίπε Γκονσάλες, πρωθυπουργός στην Ισπανία και ο πρεσβευτής της Ισπανίας ήταν ο Μιράντα, ένας χριστιανοδημοκράτης. Εγώ είχα προσεκληθεί και έμεινα ένα μήνα στο Ελσαρβαδό ζώντας όπως και εσείς. <laughs> Και μέσω διάστημα αυτό έπεσε και μια βόμβα στο ξενοδοχείο μου. επασφυρητώσει διασώθηκα. Και στην πρεσβεία της Ισπανίας είχα την ευκαιρία να συναντηθώ κρυφά με τους εκπροσώπους του μετόπου Φαραμπούντι το Μαρτί για να γίνουν οι πρώτες ενέργειες οι οποίες οδήγησαν εν καιρό στην ειρήνευση. Εσείς είσαστε πια πραγματικά μια απόδειξη του πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνευση και επανενσωμάτωση όπως γίνεται τώρα η ίδια προσπάθεια στην Κολομβία. Εγώ είχα την ευκαιρία να δω την κατάσταση της πολιτικής αντιπαράθεσης που προηγήθηκε τις συμφωνίες του 1972, τη δολοφονία του Κυριακουρία, όλα αυτά τα είδα με τα μάτια μου. Είδα την ε, εκστρατεία των ουλαμών του θανάτου και τελικά παρόλα αυτά μπόρεσα να γνωρίσω και την ειρήνη στο Ελσαλβαδόρ. Υπήρξε λοιπόν μια διαδικασία ομαλοποίησης, η ανάδυση νέων πολιτικών δυνάμεων από την δεξιά, την κεντροδεξιά, υπήρξε η εναλλαγή στην εξουσία και έχουμε πια κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ίσχυε στη δεκαετία του 80 και ευτυχώς έχει εξαλειφθεί. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια αφόρητη βία στη χώρα αυτή, τη φιλική μας χώρα, όπου η κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ χάνει το κύρος της γιατί υπάρχει μια εντύπωση ότι με την μεγάλη έκταση της βίας αυτό δείχνει να υπάρχει απουσία του κράτους σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ που μπορέσατε να καταλήξετε σε αυτήν τη συνένεση για να δοθεί μια πολιτική λύση στο θέμα αυτό. Και οι πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνικοί οικονομική οικονομικοί φορείς, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει την ικανότητα μιας κυβέρνησης και μόνο. Για να βγει κανείς από αυτό το αδιέξοδο, για να μπορέσει το Σαλβαδόρ να ανακτήσει το κύρος και την αξιοπρέπεια μιας σημαντικής χώρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια συμφωνία για τα θέματα αυτά. Εκεί λοιπόν όλοι οι φίλοι της Λατινικής Αμερικής θα πρέπει να βοηθήσουν και εμείς ως Ευρωπαίοι σας θεωρούμε φίλους μας και επομένως πάντα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για να επιτύχετε σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που έχετε μπροστά σας. Δεν έχετε το δικαίωμα να αποτύχετε ενώπιον αυτής της μεγάλης πρόκλησης. Γιατί ο κόσμος περιμένει ότι τελικά το κράτος θα μπορέσει να έχει μια παρουσία στην κοινωνική ζωή, στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δεν θα υπάρχουν πια αυτές οι ελλείψεις στην, κρασική, στην καθημερινή ζωή και θα σταματήσει αυτή η βία η οποία κυλιδώνει το κύρος της χώρας σας. Γιατί η ύπαρξη αυτής της βίας ήδη είναι μια σκιά σε όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει το κράτος του Ελσαρβαδόρ και τραυματίζει την αξιοπιστία του. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα πολιτικής, πρόβλημα έλλειψης ευκαιριών, έλλειψης ανισοτήτων, αυτό το χάσμα το κοινωνικό το οποίο βλέπουμε. Εσείς φυσικά έχετε την απόλυτη κυριαρχικότητα και την απόλυτη ε, δυνατότητα επιλογής των λύσεων που θα προκρίνεται. Αλλά εμείς από τη δική μας πλευρά Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι για να επιτευχθεί μια συνένεση τέτοια έκθεση για την εξάλληψη τη ε, βία στην αγαπημένη από εμά αυτή η χώρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα στο οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να σα βοηθήσει με όλα τα μέσα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει ε, ο, ο κύριος Σι. Yes, correct. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερο στο σχέδιο ασφάλεια που μας παρουσιάσατε ότι έχετε στο επίκεντρο την πρόληψη. Είναι σημαντικό τμήμα της στρατηγικής σας η πρόληψη. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ πετυχημένη τη στρατηγική σας και το σχέδιο ασφαλείας για το Ελ Σαλβαντόρ. Πρόσφατα είδαμε ότι κάποια πολιτικά κόμματα και οργανώσεις ζήτησαν από το κράτος να επανέλθει σε μια πολιτική καταστολής ε, και πολύ αυστηρή. Πώς θα ε, αντισταθείτε σε αυτό το, ε, τον πειρασμό να επιστρέψετε σε πιο σκληρή πολιτική και καταστολής και να απομακρυνθείτε από την πρόληψη. Επίσης μιλήσετε για τη χρηματοδοτική πτυχή του σχεδίου και είπατε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα με τα δημόσια οικονομικά. Φυσικά αυτή τη στιγμή με την παγκόσμια κρίση κανένας ε, δεν ε, είναι σε καλή θέση. Αλλά μας είπατε ε, για τη χρηματοδοτική πτυχή. Ποια είναι η χρηματοδοτική ικανότητα αυτού του σχεδίου. Θα έχετε μια πιο σφαιρική προσέγγιση και σκέψη για μια προοδευτική και φορολογική μεταρρύθμιση ενδεχομένω, προκειμένου να χρηματοδοτήσετε πιο εύκολα αυτό το σχέδιο. Επίση, ε, ήδη η Oxfam συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Πώς σκοπεύετε να εντάξετε στην εφαρμογή του σχεδίου και οργανώσει κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή του σχεδίου. Και πώς θα εξασφαλίσετε ε, έλεγχο της ε, χρησιμοποίησης των κονδύλων και από εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών, Σαν να υπάρχει μια λογοδοσία. Επίσης, μιλήσαμε για μια σφαιρική αντίληψη της ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό η ασφάλεια των γυναικών έχει θεμελιώδη σημασία και είμαι μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε δύο μέρες θα έχουμε και την ε, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου. Δυστυχώς όμως στο Ελσαλβαντόρ έχουμε γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους, ε, έχουμε γυναίκες που βρίσκονται στις φυλακές, παρά τις καλές προθέσεις και επίσης πριν από λίγους μήνες προσπαθήσατε να ξεκινήσετε μία μεταρρύθμιση ώστε να συμπεριλάβετε και στα σχέδιά σας μία θεραπευτική ε, άβλωση, άβλωση για θεραπευτικούς σκοπούς. Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε και το θέμα της προστασίας της ακαιρεότητας των γυναικών στο Ελσαλβαντόρ στο σχέδιό σας. Η Βερόνικα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας, η ομιλία σας και όπως είπε και ο Λουίς Δεγκράντες, ερχόμαστε κοντά σε έναν αδελφό λαό πραγματικά. Το σχέδιό σας είναι πολύ φιλόδοξο, βέβαια το διάβασα πολύ γρήγορα, ε, είδα μόνο τις αδερές γραμμές. Θα θέλαμε μια πιο λεπτομεριακή ανάλυση, μια πιο διεξοδική παρουσίαση αυτού του σχέδιου. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας στείλετε πληροφορίες για συγκεκριμένα σχέδια, κατάλαβα ότι το σχέδιο αυτό γίνεται, εφαρμόζεται και σε συνεργασία με τη, τους Δήμους και τις τοπικές αρχές. Και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για ευάλωτες ομάδες, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα αμέσως, αλλά μια σταδιακή βελτίωση. Επίσης, περιλάβατε και στα σχέδιά σας ένα σχέδιο για την ανεργία των νέων. Και εμεί έχουμε πρόβλημα με την ανεργία των νέων, ιδιαίτερα στην Ισπανία. Έχουμε τεράστια προβλήματα με τη μάστιγα αυτή για τους νέους. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ε, ποια είναι τα δικά σας σχέδια και φυσικά θα μπορούσαν και εκπρόσωποι των εργοδοτών και των επιχειρηματιών να μας δώσουν κάποιες ε, παρατηρήσεις και κάποιες προτάσεις γιατί πολλές φορές και οι επιχειρηματίες ε, δεν προσφέρουν αρκετές θέσεις απασχόλησης. Και κάτι συγκεκριμένο, τι θα συμβεί με αυτούς που έχουν απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφουν στο Ελσαλβαδόρ, θα επιστρέψουν στο Ελσαλβαδόρ και στο Μεξικό, το ίδιο πρόβλημα μας επισήμανε οι μεξικανικές αρχές. Πώς ε, θα ξαναδεχτείτε όλους αυτούς τους απόδημους ε, του Ελσαλβαδόρ που θα επιστρέψουν αργά ή γρήγορα ε, γιατί θα πρέπει, αν έχουν κάποια καλή κατάρτιση, να αναζητήσουν μια θέση επασχόληση ή να του βοηθήσετε για μια καλύτερη κατάρτιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βερονίκη. Κυρία Αντρικιένε. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για τα επιτεύγματά σας. Μας τα παρουσίασε ο Υπουργό Εξωτερικών και εγώ, ω μέλο αντιπροσωπείας... Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικά τα επιτυγματά σας στην καταπολέμηση της βίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Σας ε, συγχαίρω και ελπίζω ε, θα δείξετε την πολιτική βούληση σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και θα λάβετε την απαραίτητη και διεθνή υποστήριξη και συνδρομή για την εφαρμογή του σχεδίου σας, προκειμένου να γίνει αυτή το συντομότερο δυνατό και να είναι εκτενής. Ε, οι, χώρες, οι γειτονικές σας χώρες είναι η Γοτεμάλα και η Ονδούρα. Στις δύο αυτές χώρες γνωρίζουμε ότι τα επίπεδα βίας ε, και εγκλήματος είναι επίσης υψηλά. Διαρωτώ με λοιπόν, προβλέπετε κάποια συνεργασία με τις γειτονικές σας χώρες στο σχέδιο ασφαλείας για το Ελσαλβαντόρ. Επίσης, μια τέτοια συνεργασία θα σας βοηθούσε στη σωστή εφαρμογή του σχεδίου σε ό,τι αφορά επίσης το σχέδιο, το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, ξέρω ότι θα υποστηρίξουν και τα Ηνωμένα Έθνη την εφαρμογή του σχεδίου. Ε, εμπράκτος ε, πώς ε, διαμορφώνεται αυτή η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ. Ο Κάρλος Ζωγίνιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για την παρουσία, που μας κάνανε, να χαιρετήσω την ε, δημιουργία αυτού του σχεδίου για το ασφαλές Ελσαλβαδόρ. Πρόκειται για μια συνολική, μια παγκόσμια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε αντιπαράθεση σε πολλές χώρες του κόσμου σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές φορές σε υπηρετικό ή σε πλανητικό επίπεδο, να τροποποιήσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και η αντιπαράθεση να γίνει κοινή συναντήληψη, κατανόηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ένα σχέδιο που εξασφαλίζει την ασφάλεια χωρίς μια πραγματική συνεργασία, χωρίς ένα αγώνα κατά της ένδυας και ένα αγώνα κατά της ανισότητας. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος τρόμος για να μπορέσει να υπάρξει η ασφάλεια και η ύπαρξη ασφάλειας σε μια περιοχή είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει κανείς και τις ροές που προκαλούνται, προξενούνται από την ανασφάλεια και μεταφέρουν το πρόβλημα σε άλλα εδάφη. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω την επιτυχία σας στην εκπόνηση και στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου και να τονίσω ότι η συνεργασία του Ελσαλβατόρ με τις όμορες χώρες του και με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε την ειρήνη και την ασφάλεια. Η κυρία Κάρολα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Και εγώ θέλω να σας ε, ε υποδεχθώ με εγκαρδιότητα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να τονίσω το μεγάλο σεβασμό που νιώθω για σας, για την όχι και τόσο εύκολη κατάσταση που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρατε, γιατί δώσατε έμφαση στην εκπαίδευση ως όχι μόνο προετοιμασία για την εργασία, αλλά και σαν τρόπο να ξεπεραστούν τα κοινωνικά χάσματα και έτσι να υπάρξει και κοινωνική συνένεση. Ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα αν έχετε κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές ενέργειες τις οποίες έχετε σκοπό να προβείτε σε αυτές. Δεύτερον, ποια είναι η κατάσταση των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ελ μπορείτε να μας παρουσιάσετε την τωρινή κατάσταση ίσως. Και τρίτον, με ποιο τρόπο θα συμπεριληφθεί η κοινωνία των πολιτών στο σχέδιό σας Ποιε θα είναι οι δυνατότητε να είναι ενεργή η κοινωνία των πολιτών σε αυτό το σχέδιο. Θέλω να τονίσω σίγουρα το ότι σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει αυτό το σχέδιο, ώστε να μην είμαστε αδρανείς παρατηρητέ, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και αρρωγοί και έτσι να μπορέσουμε να βρούμε τι δυνατότητε για να κάνουμε πιο εύκολο το έργο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Σέντερ. Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτού του σχεδίου και κυρίως να σας ευχηθούμε ε, συνέχιση αυτής της επιτυχίας. Γιατί αισθανόμαστε αδερφοσύνη σε τέτοιες φάσεις ε, όταν βλέπουμε ε, πώς έχετε ξεκινήσει και έχετε μπει στο καλό δρόμο Θέλω να ρωτήσω αν ε, μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κεντρική Αμερική υπάρχει κάτι πολιτικός πυλώνας, οικονομικός πυλώνας που να μπορέσει να βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να βελτιώσουμε με τι θα μπορεί να μας πει η Κομισιόν λοιπόν για να στηρίξουμε περισσότερο αυτές τις δράσεις και τις δραστηριότητες μέσω και μακροπρόθεσμα που έχετε επιτάπητες, γιατί αυτό θα αποδείκνει κιόλας ότι η συμφωνία της Λατινικής, με τη Λατινική Αμερική δεν είναι απλά μια εμπορική συμφωνία που είναι σημαντική, ναι μεν, αλλά ε, είναι μια συμφωνία που περιλαμβάνει πολιτικές και κοινωνικές πτυχέ που είναι σημαντικές για το δρόμο τον οποίο ακολουθείτε εσεί αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν αν μπορούμε να σα βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι νομίζω σκόπιμο ναι, να δώσουμε το λόγο ε, και στον εκπρόσωπο της δράση ε, Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, και φαντάζομαι ότι οι βουλευτέ θα περιμένουν περισσότερο τι απαντήσει των ε, προσκεκλημένων σα. Ε, Εμεί πάντω ε, παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία και έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία με αυτές τις αρχές της ένταξης. Πράγματι όλοι οι φορείς συμμετέχουν ή καλούνται, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχουν στην ε, διαδικασία αυτή. Ε, ε, μιλάμε επίσης για ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με καταστολή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που προκαλούν τη βία, τη ρίζα του κακού δηλαδή, μέχρι την ένταξη των ανθρώπων που βγαίνουν από τις φυλακές και πάλι στην κοινωνία. Και ιδιαίτερα αυτή η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική για γιατί Όντω είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί το να μην υπάρχει εγκληματικότητα, αλλά ταυτόχρονα και να μην ξεπερνώνται τα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των κρατικών μηχανισμών. Αυτό που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο κύριο Ασμπούν, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα εθνικό ε, project, δεν είναι ένα κυβερνητικό project. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να υπάρξει μια συνέχεια ε, για να υπάρξουν αποτελέσματα πέρα από τα στατιστικά αποτελέσματα. Οι στόχοι είναι πολλαπλή. Αν μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο ε, δύο λεφτά το λόγο στον συνάδελφό μου που είναι τοποθετημένο στο Ελσαλβαδόρ, στον κύριο Πρέσβη, για να μας πει τι κάνουμε ήδη συμβάλλοντας σε αυτό το project. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε Χαρακή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Σακοράφα. Θα σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που μπορώ να πάρω το λόγο, έστω και σύντομα. Ήθελα να πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρακολουθεί και ε, συμβάλλει στο πρόγραμμα αυτό από την αρχή μέσω ε, διαφόρων ομάδων. Είμαστε μέσα στην τεχνική γραμματεία των δύο συμβουλίων που αναφέρθηκαν ε, και που ανέφερε και ο Υπουργό Εξωτερικών. Στηρίζουμε λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλεία. Είναι πολύ σημαντική στήριξη και από πολιτική άποψη, γιατί και τα κράτη-μέλη που είναι παρόντα στο Ελσαρβαδόρ παρουσιάζουν, ε, συμμετέχουν συγγνώμη, στο Συμβούλιο και επίσης λοιπόν στηρίζουμε αυτόν τον διάλογο των πολυμερή που δεν είναι πάντα εύκολος. Ε, ε, και προσπαθούμε όλοι ώστε να ε, επιτύχουμε συνενέσεις. Στηρίζουμε και οικονομικά τα προγράμματα αυτά μέσω των ε, διαφόρων μας αναπτυξιακών μέσων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα συνυπογράψαμε μια σύμβαση χρηματοδότησης 50 εκατομμύρων ευρώ για κοινωνικές πολιτικές του Ελσαλβαδόρ με βάση το κοινωνικό πλάνο του πρόγραμμα της χώρας και προβλέπουμε και ενίσχυση στα μέσα πρόληψης του σχεδίου για το ασφαλέ Σελβαδόρ. Είναι ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορώ ακόμα να σα ανακοινώσω νούμερα γιατί είμαστε στη διαπραγμάτευση. Πάντω είμαστε εκεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή ε, παρακολουθούμε τα πράγματα και θέλω να πω κάτι για το Ελ και για την κυβέρνηση. Το βαθμό ανοίγματο που έχει αυτή η χώρα είναι εντυπωσιακό. Είναι τιμή μου να εργάζομαι στο Συμβούλιο ασφαλεία με την κοινωνία των πολιτών με την κυβέρνηση. Ε, πραγματικά όλοι μας ε, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε που μας αφήνουν να συμμετέχουμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Προηγουμένως, ε, μία ευρωβουλευτής ρώτησε τι είδου συγκεκριμένε δράσει περιλαμβάνει το σχέδιο και ζήτησε λεπτομέρειε. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο μια μη κυβερνητική οργάνωσης και δεν, δεν έχουμε συχνά τέτοιε ευκαιρίες. Μία λοιπόν μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο δήμο θα μας εξηγήσει πώς εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο επιτόπου. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Conex Europa. Αλεχάνδρο, έχεις το λόγο. Όπως είπε και ο συμπρόεδρος Χαουρεγγί, η Conex Europe ε, εφαρμόζει ένα σχέδιο για την πρόληψη της βίας από το 2015 στο διαμέρισμα Δελγάδο σε, σε συνεργασία με ένα γειτονικό δήμο, ο Καταλσίνκε και έχουμε επικοινωνία και συνεργασία με το σχέδιο ασφαλείας του Σαλβαδόρ και με βάση τις πέντε συνιστώσεις με μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Θεωρούμε ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Σαλβαδόρ είναι επιτυχημένο γιατί ε, κατάφερε να εμπλέξει τόσους φορείς στη χώρα και μάλιστα οι επιτυχίες που έχουμε στο διαμέρισμα Δελγάδο, τα αποτελέσματα είναι εμφανέστατα και μάλιστα έχουμε πρόοδο που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητη σε ό,τι αφορά την παρουσία μας. Ε, και επίσης ε, κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό χάρη στη συμμετοχή των πολιτών στο Δήμο, στα διαμέρισμα, στο, στους Δήμους του διαμερίσματος αυτού. Επίσης, ε, γνωρίζουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τη βία ε, που έχει τεράστια κινητικότητα και περνά πολύ εύκολα από τον ένα κλάδο στον άλλο ή ε, μετα, μεταφέρεται από τι μεγάλε πόλει προ την ύπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν το σχέδιο να προσαρμόζεται στην κινητικότητα τη βία και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη βία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το θέμα του εκβιασμού που γίνεται προς τους μικροεπιχειρηματίες ή ενδοοικογενειακή βία, βία στα σχολεία πρόσβαση στους, ε, στις δημόσιες υπηρεσίες, που επίσης είναι δύσκολη πολλές φορές. Και τέλος, ναι, θα ήθελα, θα να εκφράσω μία ευχή και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την κοινότητα του Ελσαλβαδόρ να δίνει προτεραιότητα σε σχέδια όπως αυτό με τους Δήμους που είναι ελαστικά, που πηγαίνουν επί τόπου, που ε, δίνει ε, ευκαιρίες σε τοπικές κοινότητες, σε σχολεία, σε εκκλησίες, και φέρνει αυτό το σχέδιο επιτόπου σε συγκεκριμένους δήμους. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να ε, δοθεί και χρηματοδοτική συνδρομή στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί η πρόληψη αφορά όλες τις γενναίες και θα πρέπει σε αυτόν επικεντρωθούμε. Επίσης, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της εγκατάλειψης ε, του σχολείου. Να σταματήσουμε, να αναχαιτήσουμε την ε, ε, προέλαση των συμμοριών και να βοηθήσουμε τα παιδιά να παραμείνουν στα σχολεία. Σας ευχαριστώ και το λόγο. Μέχρι τις 5.30 έχει ο Υπουργός του Ελσαλβαδόρ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλια και στις ερωτήσεις και αν χρειαστώ τη βοήθεια των συναδέλφων θα τους δώσω το λόγο. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται για μια κρατική πολιτική στην οποία συμμετείχαν διάφοροι τομείς της κοινωνίας του Ελσαλβαδόρ. Γι' αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερος τα σχόλια του Ευρωβουλευτή Ντεγκράντες Πασκουάλ Δηλαδή, έγινε αντιληπτό ότι ένα πρόβλημα τέτοιων διαστάσεων δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε παρά μόνο με συνεργασία με τους διάφορους τομείς και κλάδους της ε, κοινωνίας του Σαλβαδόρ. Φυσικά έγιναν συζητήσεις ε, για το πού θα πρέπει να δώσουμε έμφαση για τις προτεραιότητες του σχεδίου και θα το διαπιστώσετε και από την παρουσίαση και από τον προπολογισμό ποιε είναι οι προτεραιότητες μας στο σχέδιο για την ασφάλεια του Σαλβαδόρ. Και φάνηκε αυτό και από το ποιου φορεί έχουμε εμπλέξει και από την κοινωνία των πολιτών και από τα διάφορου τομείς τη κοινωνία. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή μεταξύ της αυστηρής πολιτικής ε, και της πρόληψης, το Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ μια συνενετικής διαδικασία, ε, σφαιρικής ολοκληρωμένη και φυσικά ε, έχει και μια συνιστόσα καταστολής ε, και δίωξης του εγκλήματος, αλλά έχει και μια σημαντική συνιστόσα πρόληψης και εξάρθρωσης ε, των αιτίων του κακού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, φυσικά και έχουμε δυσκολίε, δεν είμαστε οι μόνοι. Πολλέ χώρε αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε, αλλά δώσαμε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτή τη συνιστόσα τη ασφάλεια. Και όπω είπε ο Άτο Μπούν, Έχουμε συγκεκριμένο κονδύλιο για τα σχέδια ασφάλειας που είναι πέραν της γενικής συζήτησης, αλλά γίνεται και γενική συζήτηση για την ανάγκη να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην συγκέντρωση κονδυλίων, στην δημιουργία εσόδων. Πάντως αυτή η βασική συνδρομή έχει κατοχυρωθεί από τα γενικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά την ανάμειξη στο σχέδιο των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό, δημοτικό και σε επίπεδο εκπόνηση αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής. Το ακούσατε και από τον εκπρόσωπο της μη κυβερνητικής οργάνωσης και το κλειδί είναι η συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εκεί η κεντρική κυβέρνηση ε, δεν, θα έχουν πια, δεν θα έχει πια τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πρέπει να αναδείξουμε και την ε, σημασία που έχουν οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες σε αυτή τη συμμετοχική διαδικασία. Επίσης, ένα πιο γενικό θέμα, η κατάσταση της χώρας και τα νομοθετικά ζητήματα. Όπως γνωρίζετε, έγινε μια πρόταση στο Κογκρέσο του Ελσαλβαδόρ για το θέμα των αμβλώσεων. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει εμβριθής συζήτηση και η κυβέρνηση ανάλογα με τις συμφωνίες που θα λάβει το Κογκρέσο θα δράσει αντίστοιχα. Πάντως είναι επιτάπητο το πρόβλημα και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις όπως γίνονται συνήθως στις Βουλές. Και η συνεργασία με τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα επίσης είναι θεμελιώδου σημασία, γιατί έχουμε το σχέδιο της συμμαχίας για την ευημερία στο Βόρειο Τρίγωνο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες συνεργασίας. Ξεκίνησε για την περιορισμό των παράνομων μεταναστευτικών ροών, αλλά επεκτάθηκε και στο ζήτημα της αντιμετώπισης της βίας, γιατί ένας από τους πυλώνες είναι η επένδυση στα θέματα της ασφάλειας. Οι κυβέρνηση των τριών χωρών, Γουατεμάλα, Οδούρα και Ελσαλβαδόρ, επένδυσαν σε αυτό το σχέδιο περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια με συγκεκριμένα κονδύλια στις επιμέρους χώρες για να βελτιωθεί ασφάλεια στα, στους, χώρους, τόπους προέλευσης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωση του επενδυτικού και εργασιακού κλίματος και εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Ζητήσαμε μια συνδρομή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2016 εγκρίθηκαν 750 εκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρικοδότηση αυτού του σχεδίου για τη Συμμαχία για την Ευημερία στο Βόρειο Τρίγωνο. Οπότε σα διαβεβαιώ ότι έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία με τι γειτονικέ χώρε, αλλά έχουμε και μια γενικότερη στρατηγική με τι χώρε τη Κεντρική Αμερική για τη στρατηγική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Αμερική. Και ευχαριστώ του πρέσβει των χωρών τη Κεντρική και Λατινική Αμερική για την παρουσία του και του απευθύνω θερμότατο χαιρετισμό. Επίσης, ό,τι αφορά τα άλλα μέτρα, στον τομέα της παιδείας, ο Άτος Μπούν ε, διατέλεσε και υπουργό ε, Παιδείας, οπότε είναι πολύ εξοικειωμένο με το θέμα των επενδύσεων στα ζητήματα της εκπαίδευσης και επίσης ε, το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και μάλιστα πλήρους απασχόληση. Θέλουμε οι σπουδαστές να μένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στα σχολεία, όχι μόνο για να παρακολουθούν το κανονικό, το βασικό σχολικό πρόγραμμα, αλλά και επιπλέον ε, επικουρικά και προαιρετικά προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, ε, εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, που είναι πολύ σημαντική. Και τώρα, ποια συνιστόσα τη Συμφωνία σύνδεση ε, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε με τέτοιου είδους προγράμματα. Έχουμε δύο πυλώνες των πολιτικό διάλογο και τον πυλώνα της συνεργασίας. Στον πολιτικό διάλογο εντάσσεται το θέμα της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί κάλλιστα θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε με το σχέδιό μας. Και επίσης ε, θα ήθελα να σας ζητήσω, να ζητήσω από τα κοινοβούλια που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής να το κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αν δεν κάνω λάθος πάνω από 15 κοινοβούλια έχουν κυρώσει το σχέδιο, αλλά οι συνιστώσει ε, πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της κύρωσης από όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης, ε, πώς θα προσαρμοστούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαινομένου τη βία και στην κινητικότητά τη, Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα προσαρμογή. Και κάθε εβδομάδα εξετάζουμε στο Εθνικό Συμβούλιο αυτά τα σχέδια, τα επιμέρους και την προσαρμογή των σχεδίων στα νέα χαρακτηριστικά του φαινομένου. Και υπάρχει δέσμευση όχι μόνο της, του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των θεσμικών φορέων υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπως είπε ο Άτο Ασμπούν, σε αυτό το θεσμικό μηχανισμό εγώ συντονίζω τους εσωτερικούς ελέγχους για να αποφευθεί οποιαδήποτε παρουσία, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί σε τέτοιου είδους καταστάσεις υπάρχει πάντα πιθανότητα ή δυνατότητα και γι' αυτό έχουμε και την Ειδική Συγγελική Αρχή για την Πρόσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εμπλέκεται, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Έχουμε καλέσει στο Εθνικό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος και άλλο μέλος του Συμβουλίου το έχουμε καλέσει για να εξακριβώσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλο, ένα άλλο ζήτημα που είναι θεμελιώδη σημασία και το επισημάνετε κι εσεί, το θέμα τη επανένταξη των παρινοστούντων στο Ελ Σαλβαντόρ. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέραν αυτών που ακούσαμε στα μέσα μαζική ενημέρωση, μέχρι στιγμή δεν είχαμε ε, θεαματική διαφορά η θεματική αύξηση του αριθμού των απελάσεων από τι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ελσαλβαδόρ, ούτε και στην Κεντρική Αμερική. Δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, παρά την αναγγελία που έγινε για τη νέα πολιτική τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση, Μέχρι στιγμής ε, αλλαγέ στην πράξη δεν έχουμε. Πάντω έχουμε προβλέψει σενάρια επανένταξη των παλινοστούντων θα κριθεί από το πόσο θα, αυξηθεί, θα αυξηθούν τα ποσοστά ε, των επιστροφών. Έχουμε ε, σημαντικά προγράμματα ε, ώστε όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο να πηγαίνουν προς τα διαμερίσματα και τις επαρχίες ε, τις αντίστοιχες και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργασία με την Γραμματεία Διακυβέρνησης κάνουμε αυτή την γεωγραφική κατανομή. Επίσης, Όσοι υπαλληνοστούν δεν έχουν ιδιαίτερε δεξιότητε, δική κατάρτιση, φροντίζουμε να επανενταχθούν αμέσω στην αγορά εργασία. Αλλά και στου επιμέρου θεσμού ή στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε συνεχής, συνεχή παροχή συμβουλών με δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές. Επίσης, το τρίτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας και μάλιστα δίνουμε ένα αρχικό κεφάλαιο στους παλινοστούδες αφού έχουν περάσει από ένα φίλτρο για να διαπιστώσουμε αν έχουν ικανότητες να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουμε όμως ένα τέτοιο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για επανένταξη στην αγορά εργασίας των παλινοστούντων. Έχουμε επίσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε όσοι θέλουν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους, είτε στα πλαίσια της επίσημης είτε της μη τυπικής παιδείας, θα μπορούν να το κάνουν. Ε, το 2016 είχαμε 2.300 περίπου παρινοστούντες, ε, ενώ το 2016 είχαμε 21.000 ε, παρινοστούντες. Γι' αυτό και θα χρειαστούμε περισσότερους πόρους, γιατί υπήρξε αυτή η αύξηση και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διεθνή συνεργασία. Αλλιώς θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος σε αυτό το θέμα της ασφάλειας, αν δεν λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των παρινοστούντων. Επίσης έχουμε ενεργοποιήσει ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα για το διπλωματικό και προξενικό μας δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπολιτών μας και να εξαντλήσουμε τα ένδικα μέσα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων πριν οποιαδήποτε εκδήλωση ε, επαναπατρισμού προς τις χώρες προέλευσης έκρινα σκόπιμα να διευκρινίσω αυτό το θέμα που ήταν πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Άτο Ασμπούν να εμβαθύνει σε κάποια θέματα που ενδεχομένως εγώ παρέλειψα για να έχει να συμπληρώσει κάτι. Εγώ φυσικά απαντώ στα ευκολότερα ερωτήματα και αφήνω τα δυσκολότερα για τον Άτο Ασμπούν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα ερωτήματά σας. Τρία στοιχεία θέλω να τονίσω που μου φαίνονται σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, πολιτικά κόμματα. Κάποια από τα πολιτικά κόμματα πράγματι ασκούν πίεση ώστε να χρησιμοποιήσουμε σιδηρά χείρα για την πάταξη της εγκληματικότητας. Αλλά το Συμβούλιο για την Ασφάλεια στο Ελσαλβαδόρ και εμείς ως κυβέρνηση δεν συμφωνούμε ούτε θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Αποφασίσαμε ότι ως κύριο στοιχείο της δράσης μας, ως κύριο άξονα πρέπει να προωθήσουμε την πρόληψη και να προσπαθήσουμε να έχουμε την απαραίτητη ισορροπία. Πήγαμε στο, <clears throat> στην Εθνοσυνέλευση της χώρας μας και παρουσιάσαμε την θέση μας και νομίζω ότι τώρα ξεπεράστηκε αυτή η αντιπαράθεση. Οπότε αυτά που σας είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας ισχύουν απόλυτα. Δεύτερον, για τον αγώνα κατά της ένδυας που ανέφερε ο κύριος Τεγκράντες Πασκουάλ και ο κύριος Ζουρίνιου. Είναι πράγματι κλειδί ο αγώνας κατά της ένδυας, αλλά κυρίως και ο αγώνας κατά της ανισότητας. Αναφέρθηκε στην αίθουσα αυτή το όνομα δύο ανθρώπων που έχουμε μεγάλο σεβασμό για αυτούς, ο Πάδε Γιαγουρία και ο πρεσβευτής ο Άλβαρες Δεμιράντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παδεωρία μας δίδαξε και ήμουν μαθητής του ότι ο αγώνας κατά της ε, ανισότητας είναι βασικό καθήκον όλων των ανθρώπων. Πετύχαμε μια οικονομική μεγέθυνση 2,3% ετησίως, βέβαια αυτό είναι ακόμα χαμηλό ποσοστό ανάπτυξη όπως είπε ο κύριος Ραφαέλ Αλλά καταφέραμε με αυτό το χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσης να μειώσουμε την ανισότητα, την οικονομική ανισότητα κατά 10% γιατί έχουμε εστιάσει τους πόρους της μεγέθυνσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής ανισότητας. Γιατί αλλιώς θα είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο θα διαιωνιζόταν. Τρίτον, ο τομέας της ε, παιδείας. Εγώ ήμουν υπουργό παιδείας στο παρελθόν και για μένα, αυτό είναι κάτι το οποίο περιέχεται και στο σχέδιο για το ασφαλές Ελ Σαλβαδόρ, είναι απαραίτητο η αρχική παιδεία στο επίπεδο του δημοτικού και του νηπιαγωγείου και η τεχνολογική εκπαίδευση να είναι οι βασικοί άξονες της ε, παιδείας. Θέσαμε λοιπόν αυτό το στόχο ώστε πάνω από 300 300.000 παιδιά ακόμα από ότι σήμερα να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σχολική εκπαίδευση πλήρους, με, με πλήρες ωράριο. Είναι λοιπόν αυτό πάρα πολύ σημαντικό για μας η παιδεία. Η αρχική λοιπόν παιδεία από τα πρώτα χρόνια του κάθε παιδιού να είναι οικουμενική σε όλο το Σαλβαδόρ, να είναι δωρεάν και οικουμενική. Το Συμβούλιο Παιδείας, όπου είναι ο κύριος Ραφαήλ το γνωρίζει αυτό. Τέλος, να χαιρετήσω τον συνάδελφό μας, ο οποίος εργάζεται στην ε, ΜΚΟ αυτή και να εξάρω τον ρόλο των ΜΚΟ στο πρόγραμμα αυτό. Είναι σημαντική αυτή η παρουσία και θα ήθελα να βρω την ευκαιρία σε αυτή την αίθουσα να σας ε, συγχαρώ και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι η παιδεία έχει κεφαλαιόδη ρόλο και πρέπει να ενισχυθεί με κάθε μέτρο. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε το κύμα βίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και νομίζω ότι έχω απαντήσει έτσι και για αυτό το σημείο και θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή με την οποία με ακούσατε και σας ευχαριστώ που μπορέσατε να αναφέρετε και το όρμα του Πάδρε στην αίθουσα αυτή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Ασμπούν, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε, για τις πληροφορίες τις τόσο σημαντικές που μας δώσετε, για τον τρόπο που δουλεύετε αλλά και για τα αποτελέσματα που έχετε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος να μπορέσουμε να συνοψίσουμε ε, όσο μπορούμε περισσότερο και με εξαντλητικό τρόπο τα όσα ακούσαμε. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εμείς θα παρακολουθούμε και θα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη δική σας προσπάθεια, ώστε τα αποτελέσματα να είναι θετικά για τον λαό σας και αλλά γενικότερα για τον λαό της κεντρι... των κρατών της Κεντρικής Αμερικής όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε όμως να συνοψίσω σε δύο, ε, σε, σε ελάχιστα που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία ακούστηκαν στη σημερινή συζήτηση. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή τη σημαντική δουλειά που, που γίνεται από διαφορετικούς φορείς, δημόσιους φορείς, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από θρησκευτικέ οργανώσεις, από πολιτικά κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών, από την εξαιρετική συνεργασία που όπως ήδη είπατε έχετε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στην χώρα σας. Ε, θα ήθελα να καταγράψω το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ανθρωποκτονίε, μα αναφέρεται τα νούμερα και είναι εντυπωσιακά πραγματικά και σε σχέση με το 2016 αλλά και το πρώτο εξάμεινο που κοντεύει το 60% από ό,τι είπατε. Ε, θέλω να σταθώ όμω στο τελευταίο που το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο αναφερθήκατε όλοι και έχει να κάνει με την πρόληψη στα θέματα της βίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δώσατε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός της εκπαίδευσης, της παιδείας που πρέπει να λαμβάνουμε όσον αφορά ε, σε αυτό το τόσο σοβαρό ε, ζήτημα. Ε, βεβαίως είναι γεγονός ότι θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να να δουλεύει πάνω σε αυτή τη διαδικασία, να, να, να προσπαθεί, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μειώσει αυτού του είδους τα, τα εγκλήματα, την ανεργία, τη φτωχοποίηση, ε, όπως είπατε θα πρέπει να επενδύει στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, να δίνει δράσεις δηλαδή διεξόδου στους πολίτες. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για όσα άκουσα σήμερα. Θέλω να σας ξαναπώ ότι θα επισκεφθούμε την χώρα σας, θα δούμε από κοντά όλα αυτά, θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάλι από καρδιάς, να ευχαριστήσω τον Συμπρόεδρο, να του ζητήσω συγγνώμη για την παρατηρία στην αρχή της, της ε, διαδικασίας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω ε, όσους είστε σήμερα σε αυτή την ε, εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you